Καλησπέρα σα. Επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνε λειτουργία. Υπάρχουν μια σειρά συνάδελφοι, εγώ, ο κύριο Τζάκομπτζιτς και άλλοι, που επιθυμούμε πολλέ φορές να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία Catch Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος μετά το τέλος των ομιλητών επειδή ήσασταν παρούσα και στη συζήτηση εάν όσοι είναι ομιλητές και είναι γραμμένοι και ξέρουν ότι σίγουρα θα μιλήσουν για ένα θέμα ασκούν και το δικαίωμα της μπλε κάρτας στερούν εκ των πραγμάτων χρόνο σε αυτούς που είναι στο catch the eye. Δεύτερον, εσείς εκεί στο Προεδρείο μπορείτε να δείτε πόσοι βουλευτές έχουν ζητήσει catch the eye και αναλόγως εάν δεν υπάρχουν να χρησιμοποιείτε την μπλε κάρτα εάν όμως υπάρχουν πολλοί ομιλητές τότε θα πρέπει να παίρνει προτεραιότητα ο αυτός που έχει ζητήσει να λειτουργήσει το catch the eye. εγώ λοιπόν σας λέω ότι για το θέμα των σκοπίων είχα ζητήσει πρώτος να μιλήσω στη διαδικασία αυτή. Just a second, please. Και το έλεγξα. Just a second, please. to finish. I'm sorry, you asked for a point of order. Yeah, I this is a point of order and I would like to raise it and I would like to give me only 10... Ναι, είναι διαδικαστικό και 10 δευτερόλεπτα χρειάζομαι. Εντάξει, 10 δευτερόλεπτα χρόνος. Μετρήστε, 10 δευτερόλεπτα. Πρώτος, well, 10 seconds please. Sir, the 10 seconds are over. I'm sorry. Πέρασαν τα 10 δευτερόλεπτα, λυπούμε, λέει η Πρόεδρος και